Έχουμε κάποια ψηφίσματα στην ημερήσια διάταξη. Are you ready? Είστε έτοιμοι. Πρώτο είναι το ψήφισμα για την δίωξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Ξεκινάμε την τροπολογία 1, δυνατάσεις της χειρός, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κύριε Μποργέτσιο, έχετε διαδικαστικό για το συγκεκριμένο ψήφισμα. Ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θυμίζω τον κανονισμό θα ήθελα να ξέρω αν η πρόεδρος προτίθεται να χαιρετήσει δημοκρατικά το σκοτσέζικο λαό που ψηφίζει αυτές τις ώρες για την ελευθερία του. Αν το, ανεξάρτητη σκοτία. Okay, um... Καλώς. Επόμενη ψηφοφορία. Τη δεύτερη τροπολογία ψηφίζουμε. Διανατάσεις χειρός. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης. Το ψήφισμα που αφορά τον Μπουρούντι και συγκεκριμένα υπόθεση του Πιέρ Κλαβέ Μπονίμπα. Κοινό ψήφισμα Επτά ομάδες υπέβαλαν την πρόταση. Ψηφίζουμε το ψήφισμα σύνολό του. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επόμενο. Παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαγκλαντές. Κοινή πρόταση ψηφίσματος. Έξι ομάδες υπέβαλαν την πρόταση. Ψηφίζουμε ταχικό κείμενο, από την παράγραφο 2, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε το ψήφισμα του σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επόμενο ψήφισμα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία και ποιε είναι οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία. Κοινή πρόταση ψηφίσματο. Πέντε ομάδε την υπέβαλαν. Ξεκινάμε τροπολογία 4. Έχουμε προφορική τροπολογία. Ο κύριος Οστρεβίσιο. Έχετε το λόγο κύριε Οστρεβίσιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Πράγματι, η τροπολογία είναι περισσότερο γλωσσική φύσεως. Αντί δύναται, θα έπρεπε να πούμε. Αντί can be, should be. Δηλαδή τονίζει ένθερμα ότι θα έπρεπε να υπάρξει πολιτική λύση αυτής της σύγκρουσης. Ρωτού συναδέλφους, υπάρχει αντίρρηση όσον αφορά την τροπολογία αυτή. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 4. Έπρεπε να ήσασταν πιο γρήγοροι, λέει η πρόεδρος. Καλώς να δω αν είσαστε 40. Όχι, μάλλον όχι. Ψηφίζουμε την τροπολογία που τροποποιήθηκε προφορικά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 2, τροπολογία 9, δυνατά της χειρός υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 με προφορική τροπολογία του κυρίου Φλέκενστάιν. Κύριε Φλέκενστάιν, έχετε το λόγο για την προφορική τροπολογία. Ναι, κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε και στη συνεννόηση με τις άλλες πολιτικές ομάδες το τέλος της παραγράφου παριθμών 10 ε, το on the ground να αντικατασταθεί από τις λέξεις ε, στην Ουκρανία, in Ukraine. Υπάρχουν αντιρρήσεις Όσον αφορά την τροπολογία, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροποποιηθήσα τροπολογία. Υπέρ. Α, ζητώ συγγνώμη, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, παράγραφος 17. Ανατάσσεως της χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε στην τροπολογία 3. τη χειρό υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας εγκρίνεται. Παράγραφος 28. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Δυνατά της χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε. Να γίνει επαλήθευση ηλεκτρονική. Ξεκινά ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Δυνατάς ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 σε δύο τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 διανομαστικής ψηφοφορίας άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Δυνατάς της χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επόμενο ψήφισμα, η αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επιδημία της έμπολα. Έχουμε κοινή πρόταση ψηφίσματος από πέντε ομάδες. Πριν ψηφίσουμε το ψήφισμα στο σύνολό του, κυρία Βάντερ Στοκ, έχει διαδικαστικό θέμα. Ορίστε. Θα ήθελα ναι, ένα διαδικαστικό για το ψήφισμα αυτό. Εχθές το βράδυ στις 8 η ώρα το πήραμε. 27 σελίδες, μόνο στα αγγλικά δεν μιλάμε όλοι αγγλικά. 27 σελίδες στα αγγλικά. Εχθές το βράδυ στις 8 η ώρα. Πώς σας φαίνεται και 12 πρέπει να ψηφίσουμε. Παρακαλώ να γραφεί στα πρακτικά. Δεν επιτρέπεται αυτή η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σημειώνεται, αλλά σχετίζεται με την προθεσμία για τις ομάδες. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του διανατάσσεως της χειρός, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στο ψήφισμα για την κατάσταση στο Ιράκ, τη Συρία και την επίθεση της ISIS και τη δίωξη των ανηλίκων. Έχουμε κοινό ψήφισμα, κοινή πρόταση ψηφίσματος πέντε ομάδων που ψηφίζουμε. Ξεκινάμε τροπολογία 3. Διανατάσσω της χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 9 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το συνολικό ψήφισμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στο ψήφισμα για την κατάσταση στη Λιβύη. Έχουμε μια κοινή πρόταση ψηφίσματος από τις πολιτικές ομάδες. Ξεκινούμε με την τροπολογία 3, διανατάσσεω της χειρός ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στο ΚΕΙ, η λογική σκέψη, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα το ψήφισμα συνολικά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο ψήφισμα για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Λάνσο, ε, θέλετε το λόγο για διαδικαστικό. Ε, μια ερώτηση έχω να κάνω σε εσά κύριε Αντιπρόεδρε. Γιατί ψηφίζουμε πρώτα το ψήφισμα μια πολιτικής ομάδας μεμονωμένη, εφόσον υπάρχει άλλο ψήφισμα ΕΛΚ, ε, ΑΛΔΕ, Συντηρητικών και Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Έχω και δεύτερη. Θέλουμε ονομαστικές κλήσεις στι σημαντικέ ψηφοφορίες. Ενώ εδώ μια πολιτική ομάδα έχει καταθέσει ψήφισμα και ζητάει παντού ονομαστική ψηφοφορία. Για ποιο λόγο αυτό. Ευχαριστώ. Mr. Lambsdorff, it's no... Το σημειώνουμε κύριε Λάμστροφ, αλλά την απάντηση την ξέρετε. Είναι διαδικαστικό το θέμα. Αριθμητικά ψηφίζονται τα ψηφίσματα. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση των κανονισμών. Άρα νομίζω ότι καλό θα ήταν να προχωρήσουμε. Έχουμε λοιπόν την πρόταση ψηφίσματος από την ομάδα της ΓΚΟΕ. Έχουμε και μία σειρά από ονομαστικές ψηφοφορίες. Σας παρακαλώ να αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Παράγραφος 1, αρχική ψηφοφορία ονομαστικά. Αρχικό κείμενο, συγγνώμη, ονομαστικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Διαδικαστικό, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα αυτά μαζί, αν μπλοκ. Αν δεν διαφωνεί κανείς. Είναι κάποιος αντίθετος προς την ιδέα αυτή. Άρα πάμε μία-μία. Παράγραφος 8. Άρχεται η ονομαστική και πάλι ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10 στο σημείο D λατινικό άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10 σημείο Ή λατινικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10 σημείο F λατινικό. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. λατινικο αρχεται ψηφοφορια Σημείο Παράγραφος 10 σημείο I λατινικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Διαδικαστικό έχουμε. Κυρία Μπερές, θέλετε το λόγο για διαδικαστικό. Ναι, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, ίσως είμαι άπειρη Διερωτώ με όμως. Με βάση ποιο άρθρο του κανονισμού προχωρούμε στην ψηφοφορία με βάση αυτή τη σειρά που επιλέξατε. Συνήθως παραλαμβάνω ότι ίσως ε, απατώμε και θα με διαψεύσετε βέβαια. Νομίζω ότι πρώτα ε, ψηφίζεται ένα ψήφισμα που αποτελεί προϊόν συμβιβασμού πολλών πολιτικών ομάδων. Αυτό ψηφίστε πρώτα συνήθως. Από ό,τι μου λένε, είναι το κανόνα 123, παράγραφος 4. Που λέει ότι ότι ναι μεν αντικαθίσταται ε, τα ψηφίσματα που έχουν καταθέσει υπογράφονται των πολιτικών ομάδων από ένα κοινό ψήφισμα αυτών των πολιτικών ομάδων, αλλά όχι τα άλλα ψηφίσματα. Περνάμε λοιπόν στο 10 Σημείο K, λατινικό, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10, σημείο M, λατινικό, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Θεολογική σκέψη ή e, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. F. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. G. Λατινικό άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. I. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε συνολικά το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην πρόταση ψηφίσματος της ομάδος των Πρασίνων. Διανατάσσω της χειρός. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πρόταση... Μα ήταν προφανές. Πρόταση ψηφίσματος από την ομάδα EFTD. τάσω στις χειρός ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και τώρα φτάνουμε στην κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν τέσσερις πολιτικές ομάδες και ξεκινούμε με την τροπολογία 5 Ονομαστικά ψηφίζουμε άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ανακασυχηρός. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ψήφι υπέρ. Ανάταση χειρός. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ανατάσσος χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εντρίνεται. Τροπολογία 10. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Δέκα ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Διανατάσσεως της χειρός ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία 4, διανατάσσεως ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και τώρα συνολικά το ψήφισμα. Ονομαστικά ψηφίζουμε άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνάμε σε ψήφισμα σύμφωνα για τον κατεξουσιοδότηση κανονισμό σε σχέση με τα νησιά Φίτζι. Ονομαστική είναι η ψηφοφορία που έχουμε. Ε, το ε, ψήφισμα είναι ένα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και περνάμε σε επεξηγήσεις ψήφου. In two minutes. Σε δύο λεπτά.